Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Καταρχήν μια ανακοίνωση. Η Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τα κείμενα τα οποία με διορθώσεις ε, υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο θα θεωρείται ότι εγκρίνονται αν μέχρι